ώστε οι χώρες να μην ακολουθούν αποκλίνουσες πολιτικές όπως την περίπτωση της Ινδίας. Θέλουμε μια πολύ ισχυρότερη εξωτερική πολιτική. Κλείνει λοιπόν η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση του κυρίου Βότσον. Συνεπής πολιτική απέναντι σε καθεστώτα κατά τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα. Έχετε το λόγο κύριε Βάτσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους κοιόδης εισηγητές. Η έκθεση έχει το όνομά μου, αλλά είναι αποτέλεσμα κοινή προσπάθειας, διακομματικής. Ένα από τα πιο σημαντικά μέσα που έχουμε στην κοινή εξωτερική πολιτική μας είναι οι κυρώσεις ή τα περιοριστικά μέτρα τα λεγόμενα. Η έκθεση αυτή λοιπόν θέλει να καταστήσει την πολιτική μας σε σχέση με τη χρήση περιοριστικών μέτρων συνεκτική. Συστήνει όλα τα εξωτερικά περιοριστικά μέτρα να, να συνδυάζονται αν θέλετε με αντίστοιχα μέτρα εις βάρος των ηγετών των χωρών αυτών όταν είναι στο εσωτερικό των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να τους αφήνουμε και ασφαλής όταν είναι στις περιοχές που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα και δεν θα έλεγα προωθεί την αξιοπιστία μας. Ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα δεν υπάρχουν μέτρα εις βάρος τους. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση απέναντι σε αυταρχικούς ηγέτες. Πρέπει οι πολιτικές μας να γίνουν πιο αναλογικές, πιο στοχευμένες και πιο ανθρώπινες. Και θα πρέπει τα νέα μέσα που μας δίδει η συνθήκη της Λισαβόνας να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η πολιτική μας να καταστεί συνεκτική. Να τους εμποδίζουμε να έχουν στα σύνορά μας, στο εσωτερικό των σύνορων μας, οικονομικά αγαθά, να τους απαγορεύουμε ε, τα ταξίδια στις χώρες μας για μη ανθρωπιστικούς λόγους και να ζητήσουμε τα κράτη-μέλη να διώκουν αυτούς που στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους συνδράμουν και ε, δεν εφαρμόζουν τις κοινωνικές, κοινοτικές πολιτικές. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Έχουν ε, δύο στα πλαίσια, ε, ζητήσει το λόγο στα πλαίσια της διαδικασίας Catch Κυρία Κόνμπερκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα έγκαιρη και εύθετη μετά τα περιοριστικά μέτρα που λάβαμε εις βάρος του Ιράν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να κρατά ανοιχτή τη συζήτηση γύρω από τα περιοριστικά μέτρα και την αποτελεσματικότητά τους. τα πλαίσια της προσπάθειας επίτευξης της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας. Ζητάμε από το Συμβούλιο να αναπτύξει ξεκάθαρα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία θα εφαρμόζονται τα περιοριστικά αυτά μέτρα. Στην περίπτωση του Ιράν, του εμπορικού αποκλεισμού, αυτό ακριβώς χρειάζεται. Δεύτερον, η έκθεση αυτή είναι ξεκάθαρη σε σχέση με την προϋπόθεση ότι οι κυρώσεις δεν θα πρέπει να βλάπτουν τον πληθυσμό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό στην περίπτωση του Ιράν. Το μόνο που θέλουμε είναι οι Ιρανοί, ο Ιρανικός λαός να μας θεωρήσει εχθρό. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω το ότι μια συνεκτική πολιτική στο εσωτερικό των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αναγκαία. Σήμερα άκουσα από έναν πανεπιστημιακό που ήρθε στην αντιπροσωπεία με το Ιράν ότι η Αυστριακή Τράπεζα του πάγωσε 900 ευρώ που είχε σε ένα λογαριασμό ενώ σε άλλες χώρες όπως στην Μάλτα το καθεστώς έχει εκατομμύρια ευρώ που δεν τα έχει παγώσει κανείς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερέρα ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά α, τις κυρώσεις. Η επιβολή κυρώσεων είναι μονομερής απόφαση. Ε, αντί να χρησιμοποιούμε την καλύτερη μέθοδο που είναι ο διάλογος, η ε, η διπλωματική διαπραγμάτευση. Μία απόφαση που στηρίζεται στην επιβολή της βούλησης των ισχυρότερων. Αυτό είναι οι κυρώσεις. Και η λογική της ε, δύναμης ε, δεν είναι σωστή. Θα πρέπει να πρετανεύσει η λογική. Νομίζω ότι η επιβολή κυρώσεων σε μια χώρα είναι σαν να υποστηρίζουμε τη μία πλευρά των αντιπαλόμενων μερών, κάτι που συνιστά ανεπίτρεπτη επέμβαση στα εσωτερικά μας χώρες. Έχουμε πολλές περιπτώσεις, θλιβερά παραδείγματα επέμβαση στα εσωτερικά μας χώρες με την επιβολή κυρώσεων. Έτσι προωθούμε συνομιλητές ε, που εξυπηρετούν ουσιαστικά ε, τις ε, συγκεκριμένες επιθυμίες μας θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη την κυρίαρχη βούληση του λαού και όχι την επιβολή έξωθεν που καθοδηγείται κυρίως από την, ε, από την εξυπηρέτηση διαφόρων συμφερόντων. Ε, δεσμευόμαστε από το Χάρτη Ηνωμένων Εθνών από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυστυχώς δεν είναι αυτή η προσέγγιση που υιοθετείται στην έκθεση. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κούκαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ χαρά σας βλέπω να προεδρεύετε κύριε Βλάσακ. Για να χρησιμοποιήσουμε επιτυχώς περιοριστικά μέτρα θα πρέπει να διευρύνουμε την συνεκτικότητα, αξιοπιστία και διαφάνεια στην επιβολή τους. Η συντονισμένη δράση απέναντι στο Ιράν και τη Συρία δείχνει ότι για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει όλα τα κρατη να εφαρμόσουν την ίδια πολιτική και ομοιόμορφες κυρώσεις ε, στα καθεστώτα αυτά. Τα περιοριστικά μέτρα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με πολύ προσεκτικό και επιφυλακτικό τρόπο. Να είμαστε προσεκτικοί και να τα χρησιμοποιούμε με τρόπο που ε, να μην βλάπτουν τον γενικό πληθυσμό ή την ανάπτυξη ε, της κοινωνίας που θέλουμε να βοηθήσουμε να εξυγχρονιστεί και να εκδημοκρατιστεί. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία ε, εκπροσώπων αυταρχικών καθεστώτων που έχουν παγώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τις κυρώσεις, ε, θα πρέπει ε, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία να, βοηθήσουν, να, να διοχετευτούν στις κοινωνίες για να βοηθήσουν την ε, ανάπτυξή τους. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μικολάσικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και εγώ. Νομίζω ότι για πρώτη φορά προεδρεύεται εδώ στην Ολομέλεια και θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. σε ό,τι αφορά την ε, ενιαία πολιτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί εναντί των καθεστώτων αυτών. Θα πρέπει σε τομείς εξωτερικής πολιτικής να είμαστε συνεπείς σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τέτοιων καθεστώτων και των εκπροσώπων του. Προκειμένου να μην μπορούν να κρυφτούν σε ευρωπαϊκούς λογαριασμούς, να μην μπορούν να κρύψουν εκεί τα μέσα της παρουσίας τους. Και ασφαλώς φυσικά να υπάρχει απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα άτομα αυτά, με εξαίρεση ανθρωπιστικών αποστολών. Χρειάζονται λοιπόν ενιαία κριτήρια. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελέσει το Ιράν όπου ήδη ψηφίζονται τέτοιες ε, ρυθμίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία Cash Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Άστον για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Θέλω να σας συγχαρώ λοιπόν και εσάς κύριε Αντιπρόεδρε για την ανάληψη της νέας σας αποστολής και να συγχαρώ και τον κύριο Βάτσον που εξελέγει ε, πρόεδρος ε, της ε, πολιτικής ομάδας των φιλελευθέρων. Συγχαρητήρια για τις νέες σας θέσεις. Λοιπόν, η έκθεση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και σας ευχαριστώ. Είμαι ευγνώμων για την προσπάθεια την οποία κάνατε και για τη βοήθεια την οποία μου δίδετε. Σκεπτόμαστε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτών των κυρώσεων και των περιοριστικών μέτρων. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω εδώ είναι ότι είναι ένα σημαντικό μέσο της εξωτερικής πολιτικής το οποίο χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η απόφαση του Συμβουλίου αποδεικνύει ακριβώς τη σημασία που τους δίδουμε. Στόχος των μέτρων αυτών είναι να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην πολιτική την οποία ακολουθεί μια χώρα συνολικά, συλλογικά ή ατομικά ή μεμονωμένα καλύτερα. Έτσι θα καλύψουμε τις εξελίξεις και οι κυρώσεις που θα λαμβάνονται, ε, θα αποφασίζεται να υπάρξουν, θα πρέπει να είναι σωστά στοχευμένες. Όπως ακριβώς λέτε, Σερ Γκράχαμ, πρέπει να είναι πολύ συνεκτικά τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε. Θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στους συγκεκριμένους στόχους και στις ενέργειες του συγκεκριμένου καθεστώτος. η ενιαία και συνεκτική ερμηνεία των μέτρων αυτών από πλευράς μας είναι απαραίτητη εφόσον θέλουμε τα μέτρα να είναι αποτελεσματικά και να πετύχουν τους στόχους μας. Και αυτό συνδέεται φυσικά και από την υιοθέτηση αντιστοίχων μέτρων και από τρίτες χώρες. Θα θέλαμε τα μέτρα τα οποία επιβάλλουμε να γίνονται κατανοητά. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε σωστά τα μέτρα αυτά και με τη χώρα την οποία στοχεύουμε και με τον πληθυσμό της χώρας αυτής. Δεν παίρνουμε τις αποφάσεις αυτές με ελαφρότητα, αλλά έχουμε πολύ συγκεκριμένους στόχους κάθε φορά. Το παράδειγμα του Ιράν, στόχος των κυρώσεων στο Ιράν, είναι να τους πείσουμε να φέρουν εις πέρα τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναλάβει υπογράφοντας τη Συμφωνία Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων και να μας πείσουν για την επιθυμία τους να έχουν ένα αποκλειστικά πολιτικό πρόγραμμα ατομικής ενέργειας. Όταν κάποιες χώρες και κάποια καθεστώτα αποτυγχάνουν σε σχέση με την επίτευξη των στόχων τους και σε σχέση με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις ή όπως βλέπουμε στη Συρία δεν είναι σε θέση να υπηρετήσουν τον λαό τους και χρησιμοποιούν, μετέρχονται βία βάρος του λαού τους, τότε οφείλουμε να αντιδράσουμε ηθικά και αυτή πρέπει να είναι η στάση της διεθνούς κοινότητας. Στόχος ακριβώς των μέτρων είναι να πετύχουμε την αλλαγή αυτή. Ελπίζουμε αυτό να γίνει κατανοητό και εδώ, να γίνει κατανοητό φυσικά από τη χώρα προορισμού και τον λαό της χώρας αυτής. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να σεβόμεθα τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες σύμφωνα με την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα δεν είναι να διευκρινίσουμε απλά την πολιτική μας, αλλά και να ακολουθήσουμε τις ε, ε, βέλτιστες των διαθεσίμων πρακτικών. Το έγγραφο το οποίο ακολουθούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε θετικά δεκτό και από την Επιτροπή Πίεση τον Ιανουάριο. και γίνεται αναφορά ε, και στην δική σας έκθεση. Στην εισαγωγή σας αναφερθήκατε στα θέματα των εμπορικών συμφερόντων, ιδιαίτερα των ηγετών και της καθεστικίας τάξης. Ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης παγώσαμε τις καταθέσεις των ηγετών της Συρίας, της Τινησίας, της Αιγύπτου κτλ. Ακόμα και αν υπάρχει μια ειρηνική μεταβατική περίοδος, το θέμα των καταθέσεων και του πλούτου στο εξωτερικό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά και θα πρέπει να μεταφερθούν τα χρήματα αυτά στην χώρα η οποία έχει αλλάξει εν τω μεταξύ. Είναι μια δύσκολη διαδικασία και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα οργανώνει ένα workshop στην Τινησία έτσι ώστε να δούμε με ποιο τρόπο θα βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να πάρουν πίσω τα χρήματα τα οποία οι προηγούμενοι ηγέτες τους είχαν βγάλει στο εξωτερικό. Τα μέτρα μας λοιπόν θα πρέπει να είναι συνεκτικά, σταθερά και οι στόχοι των περιοριστικών μέτρων θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μην αφήνουν παραθυράκια τα οποία θα βλάψουν και την αξιοπιστία και θα μας αποτρέψουν να πετύχουμε τους στόχους μας και θα πρέπει επίσης να είμαστε σε θέση να ακυρώσουμε την εφαρμογή των μέτρων αυτών όταν επιστραφούν τα αγαθά ενός λαού στη χώρα του. Αυτά λοιπόν είναι θέματα που θα συζητήσουμε πολύ τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Άστον. Σας ευχαριστώ και για τα τελικά σας σχόλια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και για τα συγχαρητήριά σας. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί μείνατε εδώ από τις 5 το απόγευμα συνέχεια είστε εδώ μαζί μας Κάνετε μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, δεν είναι πολύ εύκολο να παρακολουθεί κανείς τόση πολλή ώρα τις εργασίες μας και σας ευχαριστώ για αυτό. Λοιπόν, κλείνει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Το επόμενο θέμα είναι πλέον η έκθεση φύσας